αύριο, 3η 20 Νοεμβρίου από τις 8.30 ε, από τις 12.30 από τις 3 ε, έως τις 8 ε, και από τις 9 έως τα μεσάνυχτα. Μπορείτε να βρείτε την ημερήσια διάταξη στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς και όλους τους συνεργάτες της Προεδρίας και εδώ ολοκληρώνω τη